της 4 ης Σεπτεμβρίου 2017 και τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Τα συνοπτικά πρακτικά εγκρίνονται.